Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Κίνα. Ε, τον ε, λόγο εξ του Συμβουλίου έχει ο κύριος Κάρλ Μπίλτ. Κύριε Μπίλτ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, άλλη μια συζήτηση πολύ σημαντική Όλες αυτές οι ταραχές στην Κίνα ε, εντοπίζονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της Κίνας, στην ε, επαρχία της Σινγκιάνγκ. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει τα επεισόδια εκεί, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι συνάδελφοί σας βουλευτές. Και από το Συμβούλιο εκφράσαμε την ανησυχία μας μετά από αναφορές για το τι συμβαίνει εκεί. Ζητήσαμε εγκράτεια και από τις δύο πλευρές προκειμένου να επιληθεί να επέλθει ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης. Φυσικά αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα και λυπούμαστε ειλικρινά όχι μόνο για τις απώλειες ζώων αλλά και για τις καταστροφές που λαμβάνουν χώρα και καταδικάζουμε τους υπέτειους αυτών των καταστροφών από όπου και αν προέρχονται. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ενημερώσω κάπως γενικότερα για τη σχέση μας με την Κίνα. Μια χώρα με την οποία έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων που είναι αρκετά περίπλοκες. Όταν το 2003 αποφασίσαμε να εντάξουμε όλες αυτές τις σχέσεις σε μια ε, περιεκτική στρατηγική εταιρική σχέση, γνωρίζαμε ότι δημιουργούσαμε ένα πολύ φιλόδοξο και δύσκολο πρόγραμμα. Η περιπλοκότητα στις σχέσεις με την Κίνα βρήθηκε ευκαιριών, αλλά και προκλήσεων διαφόρων μορφών. Αυτό προσπαθούμε στις σχέσεις μας με την Κίνα είναι να έχουμε ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο εφόλης της ύλης και για όλες μας τις ανησυχίες. Και η βάση ενός τέτοιου ανοιχτού διαλόγου είναι το κοινό ενδιαφέρον που έχουμε και το κοινό μας συμφέρον για τη σφυριλάτηση της σχέσης μας και το κοινό μας συμφέρον για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Και αυτό το επιδιώκουμε με το διάλογο. Με τις πολυμερείς σχέσεις έχουμε τις αιτήσιες ε, διασκέψεις κορυφής, έχουμε και τακτικές ε, συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών, έχουμε και εντατικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά και τομεακού διαλόγου για εμπόριο και άλλα θέματα. Έχουμε και τον ετήσιο διάλογο υψηλού επίπεδου για οικονομικά θέματα και εμπόριο. Το 2007 εγκαινιάσαμε και τις διαπραγματεύσεις για την εταιρική σχέση και μια περιεκτική συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις για την περιεκτική αυτή συμφωνία εταιρικής σχέσης προχωρούν γιατί υπάρχει τεράστιο δυναμικό και στις δύο πλευρές. Είναι σαφές και δηλωμένο το συμφέρον μας ε, για την ανάπτυξη των σχέσεων μας με την Κίνα σε πολλούς κλάδους. Και αυτό προϋποθέτει και την ε, δυνατότητα ανοιχτού και ειλικρινού διαλόγου και για θέματα όπου υπάρχει διάσταση απόψεων ή ε, διαφορά αξιών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το θέμα των αντιφρονούντων, των αντιρρησιών. Αλλά έχουμε και κοινά συμφέροντα. Για παράδειγμα, την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το θέμα της ε, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά είναι κοινά μας ε, συμφέροντα. Έχουμε και την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας με την πρόκληση από τον DPIK. Έχουμε την κατάσταση στη Βυρμανία που επίσης μας ανησυχεί. Αλλά και την κατάσταση στην Αφρική, γιατί θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις ανοιχτές θαλάσσιες διόδους στο κέρας της Αφρικής. Έχουμε πολλές ανησυχίες και για τα θέματα της ανάπτυξης. Αυτά δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε όλα διεξοδικά γιατί, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Ευελπιστώ όμως ότι οι διαφορές μας θα επιληθούν ε, εύκολα, ειρηνικά και ελπίζω να έχουμε ειλικρινή διάλογο με τους Κινέζους και για τα θέματα αυτά, αλλά και για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που μας ενδιαφέρουν και για τα οποία χρειάζεται διάλογος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Εξ ονόματος της Επιτροπής, η κυρία Κάθριν Άστον, Ευχαριστώ και χαίρομαι που σας αναβλέπω. Αξιότιμα μέλη, σημάδι της σημασίας που προσδίδει το Κοινοβούλιο Στρατηγικές Σχέσεις με την Κίνα Φαίνεται, διότι στην ενακτήρια αυτή συνεδρία έχετε βάλει αυτό το θέμα από συζήτηση και χαίρομαι που μπορώ να συμβάλλω με μια σύντομη περιγραφή τη άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου τη συναδέλφου Μπενίτο Φερέρο Βάλτνερ που όπω σα είπα δυστυχώ ταξιδεύει την εβδομάδα και δεν μπορεί να παρίσταται. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στο σώμα την τεράστια πρόοδο που σημειώσαμε σχέση με την Κίνα από την πρώτη σύνοδο κορυφή που έγινε πριν από 10 χρόνια. Οι οικονομικέ και εμπορικέ σχέσει μεταμορφώθηκαν. Οι επαφέ των λαών άτομο με άτομο πολλαπλασιάστηκαν και όλο και περισσότερα θέματα συζητάμε μαζί τους. Μετά με την τελευταία συνοδοκορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα τον Μάιο, οι διαπραγματεύσει για νέα συμφωνία εταιρική συνεργασία ε, προχωρούν καλά και εταιρική σχέσεω και έχουμε πολυάριθμες συναντήσεις υψηλό επίπεδο, Όπω τον επιστρέφηκε ο πρόεδρο Βεν τον κύριο Μπαρόσο τι αρχέ του έτου, στα πλαίσια του διαλόγου ε, υψηλού επιπέδου για το εμπόριο που συμπροείδρευσα με τον ε, κύριο Βαν Σήμερα συζητάμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη χρηματοπιστωτική κρίση και την αλλαγή του κλίματος και περιφερειακά θέματα. Ταυτόχρονα έχουμε, ενδιαφερόμαστε πολλά πολύ για τα εσωτερικά τεκτενόμενα στην Κίνα. Είδαμε πολλά επιτέγματα αλλά και κάποιες εξελίξεις που δημιουργούν ανησυχίες. Η πολιτική του ανοίγματο της οικονομίας ε, οδήγησε εκατοντάδες εκατομμυρίων να φύγουν από τη φτώχεια ε, και υπάρχει σωστή προσέγγιση των στόχων της χιλιετίας. Όμως είναι τεράστια, χανής χώρα η Κίνα, με πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα και διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Η ισχύ τη στρατηγική μα εταιρική σχέση επιτρέπει επικοδομητική ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων επιθεμάτων όπου η Ευρώπη και η Κίνα αποκλίνουν. Όπω πτυχέ των εμπορικών σχέσεων ή ανθρώπινα δικαιώματα, π.χ. το Θιβέτ, που ξέρω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο πρόσφατα εκφράσαμε μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τις ταραχές του Ζινγκ Ζανγκ. εκφράσαμε τη συλληπιτήριά μας για την απώλεια ζώων, ε, τη συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καταδικάσαμε την απώλεια ζώων Καλέσαμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση και θέλ, ζητήσαμε να τεθεί τέρμα σε κάθε βιοπραγία. Ελπίζουμε να επιληθεί το πρόβλημα ειρηνικά, ε, με διάλογο, χωρί περαιτέρω αιματοχυσία. Επί σειρά ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διαβιβάσει ανησυχίε τη προ τι κινέζικε αρχέ για την κατάσταση των νοτικών μειονοτήτων στην Κίνα και να μοιραστεί με την Κίνα την επώδυνη πολλέ φορέ εμπειρία που έχει η Ευρώπη. Πώ να αντιμετωπιστούν τα αίτια τη περιθωριοποίηση, του αποκλεισμού και τη ε, διάκριση ε, που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι μειονότητε. Αξιότιμα μέλη, όλοι συμμεριζόμαστε τον κοινό στόχο μια πιο ανοιχτή και διαφανού Κίνα, που να συμμορφώνεται με ζεθεί προδιαγραφέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνεργαστούμε με την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, εντάσσουμε την Κίνα στη διεθνή κοινότητα και θα πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγική μα συνεργασία ε, μέσω επικοδομητικού διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άστον. Ε, τώρα ε, μιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ε, εξ ονόματος Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ε, ο κύριος Έλμαρ Μπροκ. Για δύο λεπτά κύριε Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Συμφωνώ επί της αρχής με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική και να χρησιμοποιήσουμε τη συνεργασία της Κίνας. Όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να διαρρήξουμε και φυσικά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη βία, είτε πρόκειται για βία κατά διαδηλωτών. Όλα αυτά φυσικά με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά θα πρέπει να να κατανοήσουμε στην περίπτωση της Κίνας ότι με τη βία του κεντρικού στα κράτους ε, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς θα επανέρχεται με τις διαφορετικές πολιτισμικές προελεύσεις ε, όλων των ε, πληθυσμών της Κίνας. Και με την μεγάλη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία θα, προκληθούν περαιτέρω προβλήματα γιατί στην κινέζικη ιστορία βλέπουμε ότι πρόκειται για μια σειρά ε, συνενώσεων και αποσχήσεων με μεγάλη βία και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο φαύλος κύκλος και θα πρέπει να δούμε ότι οι περιφέρειες είναι ανάλογες με τη συνοτική μειονότητα δεν προκαλείται όμως από εκεί απαραίτητα τρομοκρατία και υπάρχει και το Θιβέτ. Αν δεν βρούμε με τους μετριοπαθείς κάποια συμφωνία, ε, πάντα εμφανίζονται ε, νέοι εξτρεμιστές που δεν θέλουν να περιμένουν και όλα αυτά καθυστερούν την εξέβρεση λύση σε ό,τι αφορά την εξέβρεση της ταυτότητας. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν είναι σωστό να μιλάει η κινέζικη κυβέρνηση μόνο για τρομοκράτες, για επιθέσεις κατά του κράτους κτλ. Νομίζω ότι δεν πρόκειται για λύση σωστή για τη χώρα αυτή και γι' αυτό θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμάς για όλους τους λόγους που ανέφερα. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ ο κύριος Adrian Σέβεριν, εξ ονόματος της ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός της Κίνας διερωτάται γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη του ολομέλεια της νέας κοινοβουλευτικής θητείας ε, περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη την κατάσταση στην Κίνα. Η, η απάντησή μας θα πρέπει να είναι σαφής. Αυτό συμβαίνει γιατί η Κίνα είναι πολύ σημαντική για μας και όχι επειδή πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι να δώσουμε μαθήματα στην Κίνα ή να τη επιβάλλουμε τι απόψει μα για το πώ θα πρέπει να επιλύσει τα ευαίσθητα εσωτερικά τη ζητήματα. Ακριβώ επειδή η Κίνα είναι πολύ σημαντική για μα, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα γεγονότα που επηρεάζουν την εσωτερική της σταθερότητα και σε οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλειά της. Εδώ είχαμε την πολυεθνωτική παρουσία στην ε, επαρχία ΣΥΝΚΙΑΚ και τις ε, βλέψεις της κοινότητας των Ουγγούρων σε αυτονομία. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Σίγουρα, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξασφαλίζει μια αξιοπρέπεια και ασφάλεια και για τη μειονότητα αλλά και για την πλειονότητα. Τα δικαιώματα όμω των μειονοτήτων δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσχημα και δικαιολογία για αποσχιστικέ πολιτικέ και για εξτρεμιστικά μέσα προαγωγής τέτοιων πολιτικών. Και σίγουρα θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσχημα για την δολοφονία αθών πολιτών που ανήκουν στη μία ή την άλλη θρατική κοινότητα. Ζητούμε πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τα θύματα των βιαιοτήτων, αλλά θα πρέπει να δούμε τις το πολυδιάστατο χαρακτήρα αυτού του φαινομένου και να προσφέρουμε την αρρωγή μας προς την κινέζικη κυβέρνηση και κοινωνία για να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα που προβληματίζει και πολλές ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κινέζικη κυβέρνηση να απόσχει από την υπερβολική χρήση βίας. Θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε από όλους να αποφύγουν την καταστρατήγηση των ε, μειονοτήτων ή ε, να χρησιμοποιούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων ως τρόπο εξιοποίησης άλλων συμφερόντων. Για δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, πάντα επέκρινε το Κοινοβούλιο τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στον αφαντιμετώπιση των εθνικών Οι ουγούροι της περιοχής του Σινξάν υπέφεραν περισσότερο από όλους. Κυρίως ε, μετά την κατοχή του Ανατολικού Τουρκεστάν από την Κίνα το 1949. Η λαϊκή δημοκρατία λέει ότι δεν θέλει επέκταση των εδαφών της. Η ιστορία δείχνει ότι στο Ανατολικό Τουρκεστάν, στο Θιβέτ, στην Ταϊβάν, ότι επί κομμουνιστικού καθεστώτος επεδίωκε η Κίνα να κυβερνήσει και να υποτάξει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να άρει το αποκλεισμό πολύ όπλων στην Κίνα. Ο Ευρωπαίος Πρωθυπουργός, ε, υπουργός αναφέρθη, Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο πρόβλημα αυτό και τον αποκάλεσε γενοκτονία. Αλλά η λαϊκή δημοκρατία να διαμαρτύρεται για παρέμβαση εσωτερικά της χώρας ε, δείχνει απειρχιωμένη προσέγγιση. Στη Δυτική Αμερική διαμορφώνεται η οικονομία και στην Ινδία και την Κίνα. Αν μεγάλες αποφάσεις ε, διαβιβάζονται σε νανοδευτερόλεπτα από Κίνα στις Βρυξέλλες, βλέπουμε ότι έχουμε γίνει μια παγκόσμια κοινότητα. Και σε αυτή την κοινότητα παγκόσμια δεν υπάρχει περιθώριο για καταστολή λόγω θρησκείας, εθνικότητας ή φυλής. Ε, ε, ε, δεν μπορεί να υπάρχει αντισημιτισμός ούτε φοβία του Ισλάμ. Χρειάζονται περισσότερους νέου. Έχει γεράσει ο πληθυσμό. Έχει παρόμοια προβλήματα Κίνα με αυτά που έχουμε εμείς. Το είδα όταν έκανα επίσκεψη από τέσσερα χρόνια στην Κίνα. Η λαϊκή δημοκρατία θα διαπιστώσει χρειάζεται κάποια πολιτική για την προστασία των οικονομικών μεταναστών πολιτικές για να αναγνωριστούν τα θεμητά αιτήματα των θενοτικών νεοτήτων, όπως κάνουμε και εμείς. Και εδώ, κύριε Μπίλτ, μπορεί να παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο ρημάζουν οι δημοκρατίες, τόσο πιο πρόθυμες γίνονται να επιτρέψουν αυτοδιοίκηση, αυτοκυβέρνηση ε, και το βλέπουμε και σε νεότερες ε, δημοκρατίες στην Ευρώπη, στην Ισπανία και Ουγγαρία, να βοηθήσουμε τους Κινέζους που μπορούν να ζήσουν δημοκρατικά. Το είδαμε. Είδαμε τι γίνεται στο Χονγκ Κόνγκ και στην Ταϊβάν. Και η αυξανόμενη οικονομική δύναμη θα πρέπει να ταιριάξει με πολιτική ορίμανση και θα πρέπει να διαμορφωθούν ιδέωσες πολιτικές. Πολιτικές όπως το Erasmus Mundus. Ε, πολιτικές που ανέφερε για ή επίτροπος για να αυξηθεί η ανταλλαγή ατόμων μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση για καλύτερη συνεργασία με την Κίνα. Εκ μέρου τη ομάδα των Πρασίνων Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η κυρία Χέλγα Τρίπελ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες ε, προεδρεύοντα. Καταδικάζω τη βία και από τις δύο πλευρές, και την πλευρά την Κινέζικη και από την πλευρά των Ουιγούρων. Και ε, λυπάμαι για άλλα τα αθώα θύματα, αλλά δεν πρόκειται για μία σύγκρουση ίσων δυνάμεων. Οι Ουιγούροι είναι 9 εκατομμύρια καταπιεσμένος λαός και βλέπω ότι πρόκειται για μία αποτυχημένη πολιτική για τις μειονότητες στην Κίνα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αρμονικές ε, συμβίωσεις των κοινοτήτων όπως ε, ισχυρίζονται οι Κινέζοι γιατί στην περιοχή Σινισάν υπάρχει ε, ελάχιστη αυτονομία όπως και στο Θιβέτ. Δεν υπάρχει ε, αυτοδιοίκηση. Και κυρίως αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη νέα γενιά. Δεν υπάρχουν ίσες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες και δικαιώματα για τους ε, Ουιγούρους. Αλλά το Κεντρικό Κόμμα της Κίνας ξέρει μόνο μία κατηγορία του εγκληματία αποσχιστεί. Οποιοςδήποτε στην Κίνα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αποσχιστής και ε, εγκληματίας. Αλλά θα πρέπει η Κίνα να καταλάβει ότι μόνο με το σεβασμό των ενωτήτων μπορεί να έχει μια ευκαιρία για την εσωτερική ειρήνη. Μόνο έτσι θα υπάρξει μια εσωτερική ειρηνική εξέλιξη και πρόοδος και αποδοχή της χώρας και μια σημαντική παρατήρηση προς την Σουηδική Προεδρία. Ναι, σωστά είπατε ότι έχουμε συμφέρον για να έχουμε μια στρατηγική συμφωνία εταιρική σχέση με την Κίνα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και το περιβάλλον, αλλά την κριτική για την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα δεν μπορούμε να τη θυσιάσουμε στο βωμό της εταιρική σχέσης αυτής. Θα πρέπει με σαφή για να μιλήσουμε για την πολιτική για, τα, για τις μειονότητες και για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ευχαριστώ κυρία Τρούπελ. Ε, εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών για 1,5 λεπτό ο κύριος Charles Τάνοκ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, για ένας ολόκληρος οι Ουιγούροι ζούσαν ε, σχεδόν μια παράλληλη ζωή με ειρηνικό τρόπο σε απομακρυσμένη περιοχή της Κίνας και πραγματα... Ε, πιστεύοντας ε, στο Ισλάμ. Βέβαια τώρα έχουν συνδεθεί ίσως με την Αλκάιντα. Η Κίνα έχει παρελθόν μη σεβασμού των μειονοτήτων και νομίζω ότι επίτηδες συνδέει τους Ιγούρους με την τρομοκρατία η ηγεμονία των Χάν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία από τους τρομοκράτες των Ουιγούρων. Μερικοί βρέθηκαν μέχρι το Γουαντάναμο, προσπάθησαν να σπείρουν το φόβο και τη βία. Και μάλιστα ε, θύματα της βίας ήταν και οι Κινέζοι Χάν. Πολύ ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Και εγώ ως φίλος της Ταϊβάν ε, είμαι υπέρ αυτής της θέσης. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια νέα πολιτική απέναντι στην Κίνα. Θεωρούμε το Ταϊβάν και την Ταϊβάν και το Θιβέτ τμήμα τη Λαϊκή Δημοκρατία τη Κίνα. Γι' αυτό που δεν είδε θα πρέπει να υποστηρίξουμε την απόσχηση τη επαρχία Ινγκιάνγκ. Ένα σημαντικό θέμα τη ε, υπόθεση αυτή είναι ότι ε, και ε, μουσουλμανικές χώρε παραδοσιακοί σύμμαχοι τη ε, Κίνα όπω το Σουδάν αναθεωρούν τι σχέσει του. Και ο Ερντογάν μίλησε για γενοκτονία για τους Ουιγούρους. Είναι κάπω ε, τραγική ηρωνία γιατί η ίδια η χώρα του αρνείται να αναγνωρίσει την ε, γενοκτονία των Αρμενίων. Ούτε οι ισχυρισμοί για τον παντουρκικό εθνικισμό είναι βάσιμοι, δεδομένου ότι συμβαίνει στην Ανατολική Τουρκία. Ε, εκ μέρους της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ε, ο κύριος Μπάστιαν Μπέλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στο Σινσιάν και εκτός του Σινσιάν ε, υπάρχουν απειλές για βία μεταξύ Ουγγόρων και Κινέζων. Και αυτό μπορεί να κλιμακωθεί. Και έχουμε και τη εθνική διάσταση της σύγκρουσης, στην οποία η χριστιανική κοινότητα καταδικάζει και καλεί για, δικαιότητα, για δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες του Σενσιάν. Αποδεικνύεται λοιπόν η... αποδεικνύεται έτσι η πολιτική της ε, κυβέρνησης. Στις 3 Ιουλίου κρατήθηκαν ε, οι Γούροι και εξακολουθούνται να κρατούνται. Η Επιτροπή, λοιπόν, Επιτροπή σας ε, καλό να επενδύτε για να εξασφαλίσετε ότι η κριτική αυτή κατάσταση στο Σινσιάν θα έχει ένα αντίβαρο. και αποτελέσει ένα αντίβαρο στην Κίνα προκειμένου να συμμετέχει αρμονικά και η κοινωνία σε αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Τώρα προχωρούμε στους ε, υπόλοιπους εγγεγραμμένους. Ε, για δύο λεπτά η κυρία Ανδρικιένα. Κύριε Προεδρεύοντα, κυρία Επίτροπε, η βία, πολλά θύματα, εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες στην Κίνα, στην εξέγερση στη Σενξά. Ήταν ησυχητικά τα μαντάτα που λάβαμε. Στο Σινγκιάνγκ μπλοκαρίστηκε το διαδίκτυο, περιορίστηκαν οι επικοινωνίες ε, με την περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έγιναν πριν στο Θιβέτ, τα πρόσφατα γεγονότα στο Ανατολικό Τουρκεστάν, στο Σινσάν, όπω αποκαλείται, πρέπει να είναι σήμα κινδύνου για την ε, κινέζικη κυβέρνηση και πώ εφαρμόζει την πολιτική τη για τι εθνοτικέ μειονότητε στην Κίνα. Το μήνυμα που στείλαν οι Αγκούροι είναι ότι αυτέ οι πολιτικέ απέτυχαν και ότι η κινέζικη κυβέρνηση αυτό θα πρέπει να το καταλάβει και να προσπαθήσει να βρει λύση. 8 εκατομμύρια είναι οι Αγκούροι στην περιοχή και πάντα διαμαρτυρόταν για την εντόπιση της οποίας ετύχαναν από την κινέζικη κυβέρνηση. Και έγιναν και επιθέσεις ρατσιστικής ε, φύσεως και δεν προστάτευσε ε, η Κίνα τους γιαγούρους από αυτές τις επιθέσεις. Και δεν έχει σχέση αυτό με την κατάποση τρομοκρατίας. Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί συνήθως η κινέζικη κυβέρνηση σαν πρόσχημα, σαν δικαιολογία για την καταστολή των γιαγουρών στο Ανατολικό Τουρκεστάν. Το ότι ο πρόεδρος Σινζάο έπρεπε να φύγει πιο νωρίς από τη σύνοδο G8 στην Ιταλία για να επιστρέψει στην Κίνα, δείχνει ότι η Κίνα, η κινέζικη κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι τα γεγονότα στην επαρχία αυτή δεν είναι απλώς ε, ένα επεισόδιο και αντί να προσπαθεί να καταστήλει τον κόσμο, θα πρέπει να εφαρμόσει θετικά μέτρα και να λάβει υπόψη τα βασικά αιτήματα των Ιαγούρων, κυρίως αν η Κίνα θέλει να δείξει οριμότητα και να δημιουργήσει μια πραγματικά αρμονική κοινωνία. Υποστηρίζω πλήρω λοιπόν τη θέση Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτή που εξέφρασε ο Προεδρεύων. Θα πρέπει και όλε οι πλευρέ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και η κυβέρνηση τη Κίνα θα πρέπει να σεβαστεί την ελευθεροτυπία, τη δικαίωμα του λόγου και τη ειρηνική διαμαρτυρία. Ευχαριστώ. Το, για δύο λεπτά, η κυρία Βερονίκ Τεκάιζερ. Η έξαρση της βίας στην αυτόνομη επαρχία του Σινγκιάν και η βία κατεστάλλει βία από την κυβέρνηση της Κίνας. Και μάλιστα επίσημα είχαμε 186 θύματα από την πλευρά των Ιγούρων, αλλά το αίμα εξακολουθεί να ρέει η Κίνα προσπαθεί να παρουσιάσει τις, τις βιότητες αυτές ως ε, απλή ε, ενδοεθνοτική ε, σύγκρουση. Ποια είναι όμως η, πραγματική πολιτική απέναντι στην επαρχία της ΙΓΙΑΚ που είναι μια δύσκολη και δύσκολα ελέγξιμη επαρχία που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και απαραίτητη για το ενεργειακό μέλλον της Κίνας. Βέβαια, στην επαρχία αυτή ε, διαβιούν πολλές ε, διαφορετικές εθνότητες κοινότητες, κυρίως ε, μουσουλμάνοι και τουρκόφωνοι σουνίτες μουσουλμάνοι. Και εδώ και δεκαετίες τη διακριτική μεταχείριση, ακούν απειλές εξαφάνισης, η ίδια τους η ταυτότητα απειλείται με εξαφάνιση και μάλιστα στη, στην δεκαετία του 80 ήταν κάπως πιο φιλελεύθερη η πολιτική της Κίνας αλλά με πρόσχημα την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 οι Κινέζοι εκμεταλλεύτηκαν ε, τι τρομοκρατικέ αυτέ ενέργειε για να διατρανώσουν το δικό του αγώνα κατά το, την τρομοκρατία και το θρησκευτικό εξτρεμισμό. Η Διεθνή Αμνηστία έκλεισε τον κόδωνα του κινδύνου. Μετά το Θιβέτ θα έχουμε την επαρχία τη Ινγιάνγκ. Και μετά την αποτυχία της ε, πολιτικής της Κίνας, οι ε, αποσχιστικές τάσεις των Ιγούρων βρίσκουν άλλους τρόπους για να διεκδικήσουν τους στόχου του. Δεν μπορεί η Κίνα να εξασφαλίσει τη συνοχή της με τίμημα ένα λουτρό αίματος. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον της να προσπίσει τις εθνοτικές μειονότητες. Άλλωστε, το σύμφωνο του 1984 την υποχρώνησε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Θα πρέπει να καταδικάσουμε την καταστολή και να ζητήσουμε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πραγματικό πρόβλημα στην Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να τολμήσουμε να υπενθυμίσουμε στη χώρα αυτή τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο λαό της και τον κίνδυνο που διατρέχει σε περίπτωση που αποκλίνει από το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων και την ευθύνη που φέρει απέναντι στην ε, παγκόσμια κοινότητα. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνει η Σουηδική Προεδρία. Ε, ο κύριος Πορέμπα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ο τρόπος της φήμωσης και της καταστολής ε, των διαδηλώσεων που όπως έγιναν στην Σιγιάνγκ δείχνει τον αυταρχικό και πολιταρχικό χαρακτήρα της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Κίνας. Ε, μέχρι στιγμής τα επίσημα θύματα είναι 180 και χιλιάδες τραυματίστηκαν. Θα πρέπει να καταδικάσουμε τη βία αυτή και τη διακριτική μεταχείριση για θρησκευτικού λόγους. Δεν θα πρέπει η βία ενός απολυταρχικού κράτους να κατευθυνθεί προς τη μειονότητα των Ουγγούρων. Άλλωστε δεν ήταν μόνο θύματα της απολυταρχική ε, κυβέρνησης. Και στην Ευρώπη οι χριστιανικές ε, κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να προσπίσουν τις χριστιανικές κοινότητες που διαμένουν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, στην Κίνα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που απειλούνται από αυτό. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την δίωξη των ανθρώπων αυτών, ε, το βασανισμό από τις κομμουνιστικές ε, αρχές της Κίνας και τη δίωξή τους. Γιατί ε, θα πρέπει η Κίνα να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία και την ανεξαθρησκεία. Γιατί η δίωξη της Εκκλησίας δεν θα αποφέρει αποτελέσματα. Παρόλο που η Κίνα προσφεύγει συστηματικά σε τέτοιες διώξεις η Κίνα θα γίνει πραγματικά σύγχρονο κράτο όταν αρχίσει να εφαρμόζει και την ανεξιθρησκεία και τι αρχέ τη ελευθερία. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ποσέλτ για δύο λεπτά. Η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει εκ νέου ότι το Συμβούλιο αποτελεί το στενέ σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε σαφέστατα σε ό,τι αφορά τα μετανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράστηκε με σαφήνεια. Από το Συμβούλιο άκουσα μόνο ότι και οι δύο πλευρές ε, καταδικάζονται λόγω των βίαιων πράξεων. Φυσικά και η βία από τους Ουιγούρους μας ε, βρίσκει αντίθετους. Αλλά όταν μια κομμουνιστική δικτατορία που δεν έμαθε τίποτα από την τελευταία σφαγή καταπιέζει με τέτοιο βίαιο τρόπο ένα ολόκληρο έθνος και με εθνοτικές ε, γενοκτονίες απειλεί το έθνος αυτό, μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά με τέτοια κινηζική προπαγάνδα την οποία κανείς δεν εξετάζει. Νομίζω ότι προφανώς καταδικάζουμε την, τις απόσχικες τάσεις των Ιουγούρων, αλλά είναι πραγματικά αποσχιστική αυτή η τάση όταν καίγεται ένα σπίτι και προσπαθώ εγώ να βγω. Είναι αποσχιστικό όταν προσπαθώ να ξεφύγω. Είναι αποσχετιστική αυτή η τάση. Όχι, είναι έκφραση της επιθυμίας για ζωή. Όταν, ε, αν έδιναν στους Ουιγούρους ένα περιθώριο, ένα χώρο για να ζήσουν στην ίδια του στην πατρίδα δεν θα υπήρχε τέτοια αποσχιστική τάση. Αυτή είναι η μοναδική μέθοδος καταπολέμησης του αποσχιστικών τάσεων. Δεν είναι χαρακτηριστικό των Ουιγούρων αυτό. Οι Ουιγούροι ένας λαός είναι όπως και οι Σουηδοί. Και πρέπει δηλαδή να υποταχθούμε σε μια τέτοια εξουσία πολύ απλά επειδή είναι μεγαλύτερη από ότι εμείς. Νομίζω ότι είναι μεγάλη υποχρέωση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τους Ιγούρους. Είχαμε το Radio Liberty στη Μόναχο στο παρελθόν και σήμερα είμαστε περήφανοι που τότε αφήσαμε να ακουστεί η φωνή της ελευθερίας και νομίζω ότι θα είμαστε εξίσου περήφανοι στο μέλλον που ήμασταν το επίκεντρο των ελεύθερων Ιγούρων και ελπίζω στο μέλλον να απολαμβάνουν όλοι οι Ιγούροι την ελευθερία αυτή. Η κυρία Γκέπχαρτ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι στην Κίνα υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα το οποίο και δεν θέλουμε να ε, καταργηθεί. Σεβόμαστε το κινέζικο σύστημα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα αυτό, αυτό το... Α, Αυτή η... ότι θα πρέπει να διασπάσουμε τον ενωτικό αυτό χαρακτήρα της Κίνας. Σας παρακαλώ, σταματήστε πια να μιλάτε και ακούστε με το ενιαίο σύστημα αυτό της Κίνας το σεβόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πολυμορφία των λαών που επικρατεί στην Κίνα δεν πρέπει και αυτή να γίνει σεβαστή. Και αυτό είναι που απαιτούμε ως σοσιαλδημοκράτες. Θέλουμε τα δικαιώματα του πολίτη, τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, η ελευθερία του ανθρώπου να γίνουν όλα αυτά σεβαστά στην Κίνα. Θέλουμε η ελευθερία του τύπου να γίνει σεβαστή. Θέλουμε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα προκειμένου να μας αναφέρουν ποια είναι η κατάσταση. Αυτά ζητάμε και λέμε επίσης με σαφήνεια το εξής προς τους συναδέλφους μας στην Κίνα ότι αναμένουμε από αυτούς αυτά που αποτελούν για μας βασική αρχή να αποτελούν και για αυτούς βασικές αρχές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και ότι αυτό που μας λένε οι πολιτικοί ας κοιτάξουμε πρώτα τα, κοινωνικά προβλήματα και μετά να λύσουμε και το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι εσφαλμένο. Το αντίστροφο πρέπει να ισχύει πρώτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά τα κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί πολύ απλά αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και γι' αυτό είμαστε πολύ απογοητευμένη, κύριε Μπίλτ για αυτά που μας είπατε γιατί από τα λόγια σας τι καταλάβαμε ας κοιτάξουμε από κοινού την οικονομική δραστηριότητα γιατί αυτό αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο και όλα τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Όχι, δεν είναι μέθοδος αυτή. Δεν είναι η μέθοδος που χρειαζόμαστε η μέθοδος που χρειαζόμαστε είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να πούμε ότι πρώτα θέλουμε μια κοινή βάση επί της οποίας μπορούμε να διαμορφώσουμε τη συνεργασία μας γιατί τη συνεργασία ασφαλώς και την επιθυμούμε αλλά όχι επί οποιαδήποτε βάσης. Μόνο επί μιας βάσης που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος ε, Ντέβα για ένα λεπτό. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τον κύριο Καλμπίλτ. Πολύ ισορροπημένη ομιλία του. Εγώ πιστεύω στα σύνορα των εθνών κρατών, πώς αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Και είμαι αντίθετο στη βία την αποσχιστική, οπουδήποτε συμβαίνει. Στη Σρι Λάγκα, στην Ινδονησία, στην Σρι που γεννήθηκα, στη Βόρεια Ιρλανδία όπου βάλαν βόμβες, Ισπανία ή Κίνα. Η Κίνα είναι σημαντική ε, η Κίνα. Ε, σκοτώθηκαν 184 άνθρωποι και 1600 περίπου. Και ξεκίνησε, ξεκίνησε τα γεγονότα σε ένα ε, εργοστάσιο παιχνιδιών σκοταντών. 186 χάνοι σκοτώθηκαν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταγγείλουμε. Αν το είχαν κάνει αυτό εξωτερικέ δυνάμει, κυρίω ακρεφνεί ομάδε, θα έπρεπε να δικαστούν από Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Εάν είναι θέμα εσωτερικό, είναι θέμα της αστυνομίας ε, στην Κίνα. Είναι μικρός ο κόσμος, πρέπει να συμβιώνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καλό παράδειγμα. Να υποστηρίζουμε αποσχετικέ τάσει οπουδήποτε συμβαίνει στον κόσμο κατά του πνεύματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να προσπαθούμε να ενώσουμε την Ευρώπη και να υποστηρίζουμε τη διάλυση τη Κίνα. Αυτό οδηγεί σε συγκρούσει και σε χάο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye φοβάμαι θα πρέπει να με συμβουλεύσουν οι διερμηνείς μας για το πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά. για ένα λεπτό καθένας τέσσερις ομιλητές. Πρώτα ο κύριος ε, Σόγκορ. Είναι εδώ. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε τώρα. Θα υποστηρίξουμε την Κίνα, την Ταϊβάν, τους Ουιγούρους. Θα υπερασπίσουμε τα εκατομμύρια των Ουιγούρων. Θα ταχθούμε υπέρ της ευκολότερης και πιο συμφέρουσας οδού που είναι η οδός του εμπορίου ή θα προσπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και δούμε τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έζησαν στο Σοβιετικό ζυγό και τέτοιες εμπειρίες βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα. Θα μιλήσουμε για ουσιαστική αυτονομία, για ελευθερία έκφραση. Έχουμε πραγματική εκμετάλλευση των Ουγγούρων. Όσοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να προσπίσουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας. Αυτό είναι σαφές για μένα γιατί προέρχομαι από χώρα που είχε τέτοια εμπειρία με το κομμουνιστικό καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε θέματα σεβασμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτοδιάθεσης και αυτονομίας. Θα πρέπει εμείς να είμαστε υπόδειγμα προς μίμηση. Και αυτό ισχύει και για τις νέες χώρες της Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τις εισαγωγές και του Συμβουλίου και της Επιτροπής και ίσως να φταίει και η διερμηνία, αλλά δεν άκουσα καμία φορά τη λέξη των Ουιγούρι. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Εκατοντάδες νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα της ειρηνικής διαδήλωσης. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα δικαιώματα ε, καταπιέζονται. Ακούω φυσικά στην εισαγωγή ότι μιλήσατε για διάλογο. Αλλά αυτό που θέλω να μας πει το Συμβούλιο και η, Επιτροπή είναι ποιε είναι οι συγκεκριμένε δράσει τι οποίε βραχυπρόθεσμα θέλουν να λάβουν. Ο ε, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η συζήτηση αυτή γίνεται επί της βάσης της καθολικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στη βάση της αναγκαιότητας ε, ε, διεθνών εταιρικών σχέσεων Μιλήσαμε για, ενορμον, αρμονική ε, συνύπαρξη. Αυτό αποτελεί και σλόγγαν της ε, κυβέρνησης στην Κίνα, αλλά και την επιθυμία του λαού της Κίνας. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι δικό μας καθήκον να βοηθήσουμε τον κινέζικο λαό για την επίτευξη της, κοινωνικής, της, της αρμονικής συνύπαρξης. Για την εταιρική σχέση θα πρέπει να πούμε το εξής. Μιλώντας για τη Σιντζιάνγκ θα πρέπει να αναφέρουμε φυσικά και τους Ουιγούρους. Ωστόσο, το να τοποθετηθούμε με σαφήνεια είναι διαφορετικό από το να συγκρουστούμε. Και σε αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Για τον κύριο Πόσουλτ, μιλήσατε για αποσχιστικές τάσεις. Ξέρω ότι ξέρει τα πράγματα αυτά το κόμμα σας από τη Βαβαρία, αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο κύριος Μπρόκ, θα πρέπει να συζητάμε την συνέχιση της πολιτικής μας με την Κίνα. Κύριο Στίβενσον, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν κολοσσέο λάθος να φέρουμε την Κίνα στη συζήτηση αυτή στην ίδια κατηγορία με το Ιράν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις συζητήσεις μας για τα πρόσφατα επεισόδια και στο Ρούμιτσι. Θα πρέπει να στηριζόμαστε σε πραγματικά περιστατικά, γιατί το περιστατικό της 5ης Ιουλίου ε, προϋπόθεται μια προσχεδιασμένη επίθεση κατά του πληθυσμού Χάν στην πόλη αυτή με αυτουργού τους Ουιγούρους και μάλιστα α, κάποιοι ε, Ουιγούροι είναι φονταμεταλιστές Ισλαμιστές και ζητούν ε, απόσχεση της επαρχίας και εξαιτία ε, της βιαιότητας που χρησιμοποίησαν έχασαν τη ζωή τους 100 ε, και Κινέζοι και κυρίως Κινέζοι Χάν. Και λογικό ήταν η Κινέζικη κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τις αστυνομικές δυνάμεις για να αναχαιτήσει τη βία και τις επιθέσεις των Ουιγούρων προς τους Χάν. Τι άλλο περιμένουμε να κάνει η Κίνα. Ας στηρίξουμε λοιπόν τις επικρίσεις μας σε πραγματικά περιστατικά και όχι σε άδικες ε, ε, δηλώσεις. Κυρία Λουίση, ένα λεπτό. Νομίζω ότι η σύγκρουση εδώ παρουσιάζεται πολύ συχνά μονόπλευρα. Συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται πολύ συχνά για επιθέσεις Ουιγούρων κατά των Κινέζων και μάλιστα επιθέσεις, αφήστε με να ολοκληρώσω, επιθέσεις που έχουν ρατσιστικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, διάβασα μία συνέντευξη μιας ε, γυναίκας των Ουιγούρων που είπε «Α, τι θέλετε δηλαδή να σας ε, κυβερνήσουν οι κομμουνιστές, οι Ουιγούροι έχουν πολλά πλεονεκτήματα στην περιοχή τους. Τους επιτρέπεται να κάνουν πιο πολλά παιδιά, έχουν καλύτερες ε, ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά τον χρόνο εργασίας έναντι των ε, Χαν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε πραγματικά ποια είναι η σχέση αιτία-αιτία του. Κάποιες φορές τα προβλήματα είναι κρυμμένα και συγκαλυμμένα και δεν αρκεί μια πρώτη θεώρηση. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην υποστηρίζουμε μονόπλευρα κάποιες ε, απόψεις και να βοηθήσουμε τους Κινέζους να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Γιατί η παρουσίαση της κατάστασης όπως έγινε εδώ ήταν πολύ ε, επικίνδυνη. Γιατί η κινέζικη κυβέρνηση ε, παραδέχεται τα λάθη της. Αλλά θα πρέπει να τους βοηθήσουμε στην διαδικασία αυτή του εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ. Το, ρόλο τώρα, το, το λόγο εξ του Συμβουλίου έχει ο κύριος Μπίλτ. Κύριε Μπίλτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα αν η συζήτηση αντικατόπτυσε τον περίπλοκο χαρακτήρα των θεμάτων, ε, άλλο ζήτημα. Έχουμε τα το διαφορετικό σύστημα που έχει η Κίνα και την εξέλιξή του. Τι σημασία προσδίδουμε εμείς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε Κίνα να γίνει πιο ανοιχτή κοινωνία, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα προβλήματα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα δεν είναι μοναδική που έχει αυτά τα προβλήματα όμως, δυστυχώς. Τις τελευταίες ημέρες η εθνοτική βία που ξέσπασε στους δρόμους του Ρομτσί είναι πάντα κάτι κακό. Πρέπει να καταδικάζεται. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτούς που προσπαθούν να επιτύχουν συμφιλίωση εκεί. Σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα άλλα δικαιώματα. Ξέρουμε από τη δική μας ιστορία πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα θέματα κ. Σπιτικόφ αναφέρθηκε στην αρμονική κοινωνία, σε αυτή την έννοια. Όλοι θέλουμε να έχουμε αρμονική κοινωνία στην οποία ζούμε. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε η Κίνα να κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση. Να γίνει μια κοινωνία που θεωρείται από όλου αρμονική. Από όλου του πολίτε της Κίνας. Δεν έφτασε ακόμα εκεί η Κίνα. Λίγες κοινωνίες έχουν αυτή τη μορφή. Προφανές είναι αυτό. Να σημειώσω ότι στην αρχική παρέμβαση του κυρίου Μπροκ και του κυρίου Σεβερίν και του κυρίου Βότσον είδα ότι υπήρχαν ε, πολλά σοφά σημεία που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μελλοντικέ συζητήσει. Διότι θέλουμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας που είναι σημαντική με την Κίνα, θέλουμε να καταλάβουμε όμως και πόσο περίπλοκη είναι αυτή η σχέση και πόσο πολυδιάστατη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Μπίλτ. Φτάσαμε στο τέλος της συζητήσεως και μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης δηλώσεις Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της καταστάσεως στην Ονδούρα. Πρώτος αγορητής εκ μέλους του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός ο κύριος Μπίλτ.